Um, Happy New Year, everybody. Uh, welcome back. It's... Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλή χρονιά σε όλους. Καλωσορίσατε. Ε, ε λίγο αργήσαμε να ξεκινήσουμε, αλλά ε, τώρα πια πρέπει νομίζω να ξεκινήσουμε. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο για καθυστέρηση. Εξάλλου έχουμε και απαρτία. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αυτή η συνεδρίαση αναμεταδίδεται ε, στο διαδίκτυο εκτός από τα σημεία τα οποία είναι κυκλισμένα των θυρών. Τώρα, οι ενδείξεις οι χρονικές είναι απλώς ενδείξεις, μπορεί να αλλάξουν όλα αυτά. Τώρα θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας και αναλόγως θα το ε, προσαρμόσουμε. Έχετε αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη? Όχι. Άρα δεν έχετε αντιρρήσει, άρα μπορούμε να ε, θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται. Τώρα, ανακοινώσει του Προέδρου. Έχουμε τη συνεδρίαση της 3 η ε, Δεκεμβρίου, όπου αποφασίσαμε να ορίσουμε μόνιμους εισηγητε ω εξη Η νομική βάση θα είναι η κυρία Μίση Μακιό από το Ρενιού. μετά έχουμε τα επίμαχα θέματα. Ο κύριος Διδιέ από το ΕΛΚ, η Επιτροπολογία νομοθετικές εξουσίες ε, λοιπά. Νομίζω από τους πρασίνους, δεν ε, δεν ξέρω αν έχει επικυρωθεί. Αλλά ακόμα δεν ακούσαμε ποιο μέλος ε, θα είναι από την EOB. από το ECR, με Έχουμε για το μεταξύ ε, και περιμένουμε μέχρι την ψηφοφορία θα έχουμε τον κύριο Τουσόν από τους Πράσινους, τον κυρία Τουσάν από τους Πράσινους ε, για την Επιτροπολογία, την κυρία Σε, από το Ρινιού, όσον αφορά την άρση ασυλίας του κυρίου Άλβαρο Αμάρο, τον κύριο Χαλίκη ως εισηγητή για το αίτημα άρσης ασυλίας του κυρίου Κούναρ Μπέκ. Θα ορίσουμε τον κύριο Ιμπάν Γκαρσία Δελμπλάνκο ως εισηγητή και πρόσωπο επαφής για θέματα που αφορούν ε, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Προπολογισμού του EU μέχρι το Δεκέμβριο του 2021. Ε, έπειτα έχουμε αιτήσει για την ε, σύνταξη εκθέσεων ίδιας πρωτοβουλίας, ε, τις προκλήσεις για τους οργανωτές αθλητικών ε, εκδηλώσεων, το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Διασυνοριακών Ενώσεων και Οργανώσεων, την εταιρική δέουσα επιμέλεια και ε, ευθύνη, χρηματοδότηση των διαφορών με τα hedge funds. Τα τέσσερα πρώτα θα είναι ε, επί της ουσίας αρμόδια δική μας επιτροπή. Τώρα, έχουμε συμφωνήσει να καταθέσουμε προφορική ερώτηση για τα ε, τρισδιάστατα τυπωμένα παράνομα αντικείμενα. Αποφασίσαμε να καλέσουμε την Μαργαρέτη Φερσχάγκερ και τον Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά τη Ερή και να καλέσουμε και τον εκπρόσωπο ε, της Επιτροπής για να παρουσιάσει την έκθεση από την ε, ομάδα πυρογνωμόνων για την ε, ευθύνη και τις νέες τεχνολογίες. Έχουμε τώρα το σημείο 3 των ημερ... της ημερήσιας διάταξης, τα πρακτικά της συνεδρίασης της 3ης Δεκεμβρίου. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίας, θα θεωρήσουμε πως εγκρίνονται. Έχουμε τρία σύνολα ε, πρακτικών που δεν έχουμε εγκρίνει ακόμα για τον Νοέμβριο και πρέπει να είναι έτοιμα για την επόμενή μας συνεδρίαση. Δεν έχουμε ε, τώρα ε, επικουρικότητα στο σημείο 4, δεν έχουμε τίποτα και πάμε στο σημείο 5, κανόνες και γενικές αρχές που αφορούν μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη-μέλη και την άσκηση της Επιτροπής, ε, από πλευράς Επιτροπής των εφαρμοστικών της αρμοδιοτήτων. Ο κύριος Άγερ δεν είναι εδώ, αλλά ο κύριος Βος γενικά προσεφέρθη για να παρουσιάσει το θέμα αυτό. Οπότε παρακαλώ αν θέλετε πάρετε αμέσως το λόγο κύριε Βος. Ευχαριστώ πολύ. Εκ λοιπόν του κύριου Σάγερ που δεν μπορεί να είναι εδώ όπως είπατε και εσείς για το θέμα αυτό και μετά τις δηλώσεις Γιούνκερ όταν μίλησε για την κατάσταση της Ένωσης 14 Φεβρουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία πρόταση τροποποίησης του κανονισμού για τον κανονισμό επιτροπολογίας με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ε, που οδηγούν στην υιοθέτηση εκτελεστικών πράξεων και προτείνει σε αυτήν την ανακοίνωση Κομισιόν το σύστημα της επιτροπολογίας να παραμείνει επειδή λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά τις περισσότερες υποθέσεις, αλλά για υποθέσεις ε, ε, ευαίσθητες, ε, τα λεγόμενα opinion σενάριο, εκεί είναι πιο πολύπλοκη η κατάσταση. Ο προτινόμενο κανονισμός σχεδιάστηκε για να ταποκριθεί σε προβληματικές τέτοιες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και δραστικές ουσίες, συγκεκριμένα την γλυφοζάτη. Οπότε και δεν υπήρξε ποτέ ειδική πλειοψηφία πλειοψηφία μεταξύ των κρατών μελών που να είναι υπέρ κατά της έγκρισης ε, της γλυφοζάτης ή μεταλλαγμένων. Άρα έχουμε μη γνωμοδότηση ως αποτέλεσμα έτσι όπω είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα με τη διαδικασία επιτροπολογία, αν δεν υπάρχει υπέρ ή κατά πλειοψηφία υπέρ ή κατά τη πρόταση, ε, αν λοιπόν έχουμε μη γνωμοδότηση, η Κομισιόν μπορεί να εγκρίνει ε, το σχέδιο εκτελεστική πράξη ή να αποφασίσει να μην εγκρίνει εκτελεστική πράξη με βάση την αιτιολογία τη πρόταση. Και ενώ υπάρχει εξουσιοδότηση για την Κομισιόν να πάρει σχετική απόφαση, θεωρεί ότι παρόλα αυτά τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν τι ευθύνε του και στη συγκεκριμένη περίπτωση, επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αλλαγές στον κανονισμό περί επιτροπολογίας ε, με στόχο μεταξύ άλλων τη μείωση ε, του κινδύνου να έχουμε αυτό το σενάριο μη γνωμοδότηση, no opinion σενάριο. Παραδείγματο χάρη, προτείνει αλλαγή στου κανόνε εκλογή ε, για να μειωθεί η δυνατότητα αποχή σε περίπτωση υπουργικών διασκέψεων να δημοσιοποιούνται επίσης ψηφο, τα αποτέλεσματα των ψηφοφοριών και επίσης να υπάρχει δυνατότητα ε, να επιληφθεί το Συμβούλιο Σχετικών Υποθέσεων. Ε, ε, πέντε επιτροπές, ΑΦΚΟ, ΙΤΡΕ, ΙΝΤΑ, ΕΝΒΙ και ΕΚΟΝ έχουν γνωμοδοτήσει στο πλαίσιο της διαδικασίας συζήτηση στο Κοινοβούλιο και στις γνωμοδοτήσεις τους περισσότερες λένε ότι θα πρέπει να παραμείνει ως έχει το πλαίσιο επιτροπολογίας εφόσον λειτουργεί σωστά αλλά προτείνουν να ενισχυθεί περαιτέρω η πτυχή της ε, διαφάνειας. Το Συμβούλιο έχει υπάρξει προς το παρόν αδιέξοδο 2 Μαρτίου του 2018. Η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου έκανε μια αρνητική ε, γνωμοδότηση με βάση αυτόν τον κανονισμό και τώρα με βάση τοποθέτηση του Συμβουλίου προτινόμενος κανονισμός ε, φαίνεται να αντιβαίνει την αρχή της θεσμικής διοργανικής ισορροπίας και ε, επίσης αντιβαίνει και μπαίνει στο πεδίο των εθνικών αρχών, των κρατών μελών. Είναι προβληματική λοιπόν η οθέτηση αυτής της πρότασης ε, με βάση αυτά. Thank you for that <laughs> Εξαιρετικά τα διαβάσατε, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν ε, συνάδελφοι που θα το λόγο. Ναι, θα έρθει και η σειρά σας. Καταρχάς, να σας πω και εγώ ε, τις καλύτερες ευχές για το νέο έτος. Η κυρία Μπετίνα Μπόλαθ δεν μπορούσε να είναι σήμερα στην Επιτροπή, γιατί ταυτόχρονα συνδράζει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αλλά έχω και εγώ να διαβάσω ε, τη δική της ε, σημείωση. σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση διαδικασία επιτροπολογία. Πρόκειται για κάτι το οποίο δεν ολοκληρώθηκε στην προηγούμενη θητεία. Ο κανονισμό ε, ε, βασίζεται σε μηχανισμού ελέγχου των κρατών μελών για την άσκηση των εκκληστικών εξουσιών τη Κομισιόν. Με βάση τον κανονισμό όπω ισχύει σε περιπτώσει όπου δεν υπάρχει γνωμοδότηση από τι δύο αρμόδιες επιτροχές λόγω έλλειψης ε, ειδική πλειοψηφία από τα κράτη-μέλη, Κομισιόν ε, πρέπει να λάβει μια απόφαση εξουσιοδότηση. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί η απόφαση της Κομισιόν δεν στηρίζεται, δεν έχει πολιτική υποστήριξη. Αυτές οι αποφάσεις πολλές φορές όμως επηρεάζουν άμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες και οι επιχειρήσεις ευρωπαϊκές. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για γενετικώς μεταλλαγμένα προντέιτη γλυφοσάτη στον τομέα των τροφίμων, το Συμβούλιο μέχρι στιγμής δεν έχει εγκρίνει τη γενική προσέγγιση του επί του θέματος λόγω και της πολιτικής ευαισθησίας της σχετικής αναθεώρησης. Τώρα είναι πολύ θετικό το ότι ξεκινάνε οι συζητήσει, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, για να συνεχίσουμε το έργο μα. Βέβαια, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να μην εκπέμψουμε δηλαδή προ τα έξω λάθο μηνύματα. Πρέπει να καταστήσουμε σαφέ ότι δεν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το οποίο ε, μπλοκάρει την αναθεώρηση, αλλά τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και απευθύνουμε έκκληση στο Συμβούλιο να επιταχύνει το έργο του, το σημαντικό αυτού φακέλου, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο. Κυρία Βόλαθ, ε, βλέπει θετικά την πρόταση Κομισιόν για βελτίωση της θετικής λήψης αποφάσεων. Οι κανόνες πρέπει να αλλάξουν για να μειωθεί ο κίνδυνος του λεγόμενου no opinion σενάριο σε επιτροπές. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν να μην δονται μόνο αυτά που συμμετέχουν για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ειδική πλειοψηφία. Αν δεν υπάρχει γνωμοδότηση, θα πρέπει να υπάρχει μια άλλη δυνατότητα, δηλαδή η Επιτροπή Εφέσεων Προσφυγών να μπορεί να επιληφθεί για να έχουν και για διάφορες πολιτικά ευαίσθητες αποφάσεις ε, ευθύνη τα κράτη-μέλη. Πλειοψηφίες τώρα που γίνονται στην Επιτροπή ε, Προσφυγών θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Έτσι, να υπάρχει διαφάνεια, θα αναλάβουν έτσι ευθύνε τα κρατημέλη και θα έχουν λογοδοσία. Τελικά, ο στόχο μα πρέπει να είναι βελτίωση τη διαδικασία αποφάσεων. Άρα, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Μόνο εάν υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, θα μπορέσουμε να κάνουν τα κρατημέλη να αναλάβουν τι ευθύνε του, να λογοδοτούν περισσότερε αποφάσει που λαμβάνουν. Υπάρχει επίση δικαίωμα κοινοβουλευτική εποπτείας. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να ενισχυθεί στο πλαίσιο τη διαδικασία επιτροπολογίας. Κύριε Μπόλα, θα συναδελφός μας θα συνεργαστεί με τον κύριο Σάγερ, δεν ξέρω αν προφέρω καλά το όνομά του, και τους άλλους κοιόδης ε, και ελπίζει να λεφθεί υπόψη ε, η δική της άποψη την έκθεση του κύριου Σάγερ. Θα μπορέσουμε και την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια να συζητήσουμε αυτό το θέμα γιατί προβλέπεται δήλωση σχετική από την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να προσθεθεί στα πρακτικά, έτσι. Γίνεται. Σας το δώσω. Ωραία. Ωραία, ευχαριστούμε. ευχαριστώ. Εγώ θα είμαι λιγότερο επίσημος, δεν θα ζητήσω η παρέμβασή μου να προσθεθεί στα πρακτικά. Απλώς, κοιτάξτε, Άκουσα τον κύριο Βος και ήταν ξεκάθαρος. Και αυτή είναι μια αναπροσώνα, ένα θετικό. Ξέρω δεν είσαστε εσείς υπεύθυνο για την έκθεση. Πάντως η παρέμβαση αυτή σημειώνει δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι δεν είναι σωστό ότι όλα πηγαίνουν καλά. Όντω δεν πηγαίνουν όλα καλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν με τι άλλο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υφίσταται την ε, δηλία κάποιων χωρών μελών που προτιμούν να μην πηγαίνουν στην ψηφοφορία για να μην επιτρέψουν να δημιουργηθεί μια ειδική ε, πλειοψηφία. Συνηθίζεται αυτό σε πολλά κοινοβούλια, όχι σε εμά. Βλέπουμε όμω ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάζεται να καταλήξει σε μια πολιτική απόφαση όταν πρόκειται για τα γενετικά τροποποιημένα, για την υγεία, για θέματα πολύ σημαντικά για του πολίτε, επειδή το Συμβούλιο από τη δικιά του την πλευρά δεν θέλει να αναλάβει τι ευθύνε του. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου είναι υποχρεωμένο να προβάλλει ένσταση. Οπότε δεν είναι καλό το να είμαστε συνέχεια υποχρεωμένοι να μπλοκάρουμε τα πράγματα. Συνήθως το κοινοβούλιο υπάρχει για να δημιουργεί, όχι για να καταστρέφει. Οπότε η κατάσταση δεν είναι υπέροχη καθόλου. Για μερικά ζητήματα η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή και πρέπει να αλλάξει. Νομίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή, η οποία μπορεί να μην μπορεί να το πει, αλλά εμεί μπορούμε, ε, πιστεύουμε κι εμεί λοιπόν ότι η Επιτροπή έχει βαρεθεί και α μην το λέει. Ότι έχει από μια ε, το Συμβούλιο που δεν κάνει τίποτα και από την άλλη μεριά έχουν κάποιου άλλου οι οποίοι λένε Μα δεν έχετε δικαίωμα να μην δώσετε άδεια εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη άποψη από το Συμβούλιο και τα βάζουν με την Επιτροπή. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Η πρόταση της Κομισιόν δεν φτάνει γιατί παραμένει σε μια λογική η οποία βάζει άλλο ένα στρώμα. Δηλαδή δημιουργεί ένα τρίτο βαθμό ε, έφεσης κατά κάποιο τρόπο. Όσο παραμένουμε λοιπόν σε αυτή τη λογική η οποία λέει ότι εμείς πρέπει να παραμείνουμε σε υπουργικό επίπεδο, ίσως και σε παραπάνω επίπεδο κτλ, τίποτα δεν θα γίνει. Και εκεί όπου διαφωνώ σε σχέση με αυτά που έγιναν στην προηγούμενη θητεία και σε σχέση με αυτά τα οποία άκουσα σήμερα είναι το εξής δεν είναι δυνατόν το Συμβούλιο να μην θέλει να αλλάξει κάτι. Γιατί ναι, είναι το Συμβούλιο αυτό που μπλοκάρει τα πράγματα. Όταν λοιπόν περιμένουμε το Συμβούλιο να συμφωνήσει για να αλλάξει μια κατάσταση που το ίδιο έχει δημιουργήσει, καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύουμε να περιμένουμε επάπειρο. Γι' αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό και είχαμε επιμείνει να επανέλθει στη θητεία αυτή το ζήτημα. Είχαμε την απόφαση της ΑΦΚΟ, εγώ ήμουνα εισηγητής, οπότε υπάρχει γνωμοδότηση της ΑΦΚΟ, είναι γνωστή, έχει δημοσιευθεί. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν και είναι πολύ σημαντικό. Αντίθετα με αυτά που άκουσα, είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανεξάρτητα από τη βούληση του Συμβουλίου να μην μετακινηθεί. Αντίθετα, να δείξουμε στο Συμβούλιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει και επιθυμεί να δίνει συνέχεια, να υπάρχει διαφάνεια βέβαια μεγαλύτερη, και αυτό το λέω τόσο για την Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο. Σήμερα βέβαια δεν πρόκειται να διακανονιστεί το θέμα των πλειοψηφών κλπ. Αυτό θα συζητηθεί μεταξύ των σχεδόν εισηγητών. Αλλά επιμένω πάντως να μην φτάνει να λέμε επειδή το Συμβούλιο μπλοκάρει, επειδή η κατάσταση δεν είναι τραγική, να μην το πράγμα τόσο έχουν. Όχι, πρέπει να εξελιχθούμε και πρέπει και το Συμβούλιο να το καταλάβει. Και σίγουρα αυτό είναι το πιο σημαντικό στην απόφασή μας. Θα πρέπει το Συμβούλιο να καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με τέτοια παθητικότητα όπως το έκανε μέχρι τώρα με θέματα τα οποία δεν βγαίνουν προς τα έξω, δεν δημοσιεύονται, με χώρες οι οποίες απουσιάζουν ε, αποφασίζουν ε, με τρόπο σκοτεινό, αυτά δεν αποτελούν χαρακτηριστικά μια σύγχρονη δημοκρατίας. Εμείς θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι όλο και περισσότερο δημοκρατική. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ω νομοθέτες να ε, δουλεύουμε με κρυφές διαδικασίες και με κλειστές θύρες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριο Λεμπρετό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα εύχομαι καλή χρονιά σε όλου σα. Σήμερα συζητάμε για εκτελεστικέ πράξει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσο έχουν τα πράγματα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τι υιοθετήσει μετά από γνωμοδότηση μια επιτροπή και ενδεχομένω και μετά από μια επιτροπή που λειτουργεί μετά από έφεση. Πολύ συχνά οι επιτροπέ αυτέ όμω δεν μπορούν να γνωμοδοτήσουν, γιατί χρειάζεται δική πλειοψηφία προκειμένου να καταλήξουν σε γνωμοδότηση, είτε υπέρ είτε κατά. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα ε, όπως το βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξού και η σημερινή πρόταση. Όμως οφείλω να πω ότι εάν ε, το πρόβλημα υπάρχει, οι λύσεις που προτείνονται ε, από την άλλη δεν είναι κατάλληλες κατά τη γνώμη μου και γι' αυτό συμφωνώ αρκετά με την θέση που παρουσίασε ο κύριος Φως. Και ποιες είναι αυτές οι δύο προτάσεις. Η μία λέει ότι πρέπει να θεωρήσουμε πως για να υπολογιστεί η ειδική πλειοψηφία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μόνο τις χώρες που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, δηλαδή που δεν ε, κρατούν θέση αποχής. Την απουσία και την αποχή δηλαδή να τα αποκλείσουμε από την λήψη αποφάσεων. Κάτι το οποίο είναι κατάλληλο κατά τη γνώμη μου. Και έπειτα έρχεται και σε αντίθεση με τα προνόμια των χωρών μελών που μπορούν να αποφασίσουν να απουσιάσουν ή να κρατήσουν θέση αποχής. Και δεν βλέπω γιατί να υπάρχει τέτοιου είδου κύρωση για χώρε που έχουν την ελευθερία να υιοθετήσουν τέτοιες στάσεις. Δεύτερον, προτείνεται ενδεχομένω να υπάρξει ένας τρίτος βαθμός υποβολής ε, που να είναι στο Συμβούλιο αυτό καθεαυτό, αυτό, το οποίο θα μπορούσε να γνωμοδοτήσει απευθείας. Εδώ βλέπω ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα όμως. Κατά τη γνώμη μου, ίσως να μην κατάλαβα βέβαια καλά ποιο είναι το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για μένα το Συμβούλιο βρίσκεται πάνω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι πίστευα εγώ πάντα. Ενώ η πρόταση εδώ αντιστρέφει αυτή την ιεραρχία. Διότι καταλάβατε, το Συμβούλιο θα γνωμοδοτεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν κατάλαβα καλά, θα μπορεί να μην ακολουθήσει αυτή την γνωμοδότηση. Εδώ εγώ λέω όχι. Φέρουμε τα πάνω κάτω έτσι. Δεν είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλω εγώ και δεν νομίζω ότι είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που επιθυμούν οι, λαοί της Ευρώπης. Γι' αυτό, αν παραμείνει μια τέτοια πρόταση, εγώ θα την καταψηφίσω. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μετά από αυτό που είπε ο κύριο Λεμπρετών, θέλω και εγώ να πω ότι για να ξέρουμε ποια Ευρώπη θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, πρέπει να γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες τι συμβαίνει στου διαδρόμου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η πρόταση αυτή, ακριβώς αυτό το ρόλο έχει να βοηθήσει να υπάρξει διαφάνεια και να μπορούν αυτοί που αποφασίζουν να λογοδοτούν, να είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αυτή την αλλαγή που μέχρι τώρα υποστήριζε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν μη τι άλλο, και που τώρα υπενθύμησε και ο Πασκάλζαν. Τώρα εγώ δεν κατάλαβα ότι εδώ επανερχόμαστε στο περιεχόμενο της μεταρρύθμισης. Αυτό όμως που θέλω να υπογραμμίσω, να ζητήσω αν μη τι άλλο, είναι να δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμά μας, πώς μπορούμε μαζί να κινητοποιήσουμε τις άλλες πολιτικές ομάδες και το Συμβούλιο για να προχωρήσω αυτό το θέμα. Θα υπάρξει συζήτηση στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα και ελπίζω να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε σήμερα. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ο κύριος Φως, ευχαριστώ πολύ. Στα γερμανικά Νομίζω ότι έχουν δει και από τις ουσίες όλοι προλαλήσαντες. Το θέμα εδώ είναι πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με ρεαλιστικό τρόπο. Όταν έχουμε αυτό το αδιέξοδο από το Συμβούλιο, ε, δεν θα μπορέσουμε ίσως ε, να ε, το λύσουμε το πρόβλημα, όπως έγινε και στο τέλος προηγούμενης θητείας. Δύο λύσεις βλέπω. Το πρώτο είναι και την προηγούμενη χρονιά ο εισηγητής, ε, γιατί ήθελε η Κομισιόν απόσυρση και, μιας νέας, ε, και διαμόρφωση μιας νέας διαδικασίας. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, αν το Συμβούλιο ε, με κάποια άλλη συμφωνία ε, καταφέρει να ακολουθήσει το, το Κοινοβουλίο. Αυτό δεν το βλέπω προς το παρόν ως προοπτική. Δεν ξέρω τι γίνεται, ε, τι αποφασίζει ΑΦΚΟ και τι δυνατότητες υπάρχουν. Καλό θα ήταν αν ε, μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Αλλά το θέμα είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με κάποιο τρόπο. Εγώ δεν ξέρω τι είναι το πιο ρεαλιστικό. με κάποιο τρόπο πρέπει να λυθεί το έξοδο, θεωρώ. Δηλαδή, απόσυρση τη πρόταση και ατύπωση μια πρόταση ή μετακίνηση του Συμβουλίου. Αλλιώ δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ε, προς το παρόν δεν βλέπω κάποια άλλη εναλλακτική. Ευχαριστούμε. Θέλετε να επανέλθετε. Ναι. Κάτι που ξέχασα. Αντίθετα με τον κύριο Φως, εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Θα ήθελα, το ελπίζω τουλάχιστον και από εμά εξαρτάται, να προχωρήσει αυτή η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία τα οποία ε, ήταν θετικά, στις ακροάσεις που είχαμε με τους τωρινούς επιτρόπους ήταν και ο κύριος Σάφκοβιτς, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει διαφάνεια για πολλά θέματα. Μπορούμε να τον πιστέψουμε λοιπόν, να τον καλέσουμε εδώ, ανάλογα με το τι συζήτηση θα γίνει στην ε, Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα και μπορούμε και να τον καλέσουμε να έρθει στην Επιτροπή μας να μας πει πώς πιστεύει ότι μπορεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Πιστεύω ότι είναι σύμμαχός μας. Είναι μια πολιτική συμμαχία που χρειάζεται. Δεν πρέπει να παρετηθούμε. Σίγουρα θα πάμε πίσω αν θέλουμε την πλήρη αλλαγή, εδώ κάνουμε μερικά βήματα προς τα μπρος και πρέπει να μείνουμε σε αυτή την προσπάθεια αντί να επιμένουμε να τα ξεκινήσουμε όλα αυτού και από την αρχή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να επιθυμεί το λόγο. Δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως έχει κάτι να πει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Θα είμαι σύντομη. Το πλαίσιο της πρότασης έχει εξηγηθεί σαφώς. Το πλαίσιο επιτροπολογίας πιστεύουμε ότι πραγματικά λειτουργεί καλά. Είναι ένας ειδικό τομέας ε, αυτός που ε, στοχεύουμε με τροπολογίες εξαιτίας των προβλημάτων που έχουμε διαπιστώσει μέχρι τώρα. Που είναι περιορισμένες μεν οι περιπτώσεις όπου συναντήσαμε αυτά τα προβλήματα, αλλά είναι αρκετά δύσκολες και λεπτές. Ακούσαμε τις αλλαγές που προτείνονται και είχαμε και την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε λεπτομερώς την ε, πρόταση, οπότε δεν χρειάζεται σήμερα να το ξανακάνουμε. Είδαμε πάντως ότι το Συμβούλιο είναι απρόθυμο. Περιμένουμε την επίσημη θέση βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακόμα. Επίσης γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει συζήτηση την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Εννοείται ότι περιμένουμε την ε, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, κάτι ακόμα θέλετε να προσθέσετε κύριε Βόλτς. Μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποια μηνύματα, σινιάλα που να μας κάνουν να ελπίζουμε, να πιστεύουμε ότι κάτι κάνει το Συμβούλιο. Εγώ δεν το βλέπω κάτι τέτοιο, αλλά ίσως έχετε εσείς ε, κάποια σημάδια από το Συμβούλιο που δείχνουν ότι μπορεί και να μετακινηθεί. Απάντηση, λυπούμε. Δεν έχουμε τέτοια σημάδια από πλευρά Συμβουλίου. Κύριε Ντύρο, για να απαντήσω στον κύριο Φως, δεν υπάρχει καλύτερο δείγμα από ένα ε, ψήφισμα που να εγκρίνει ο συνομοθέτη που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να κάνουμε πολιτική. Δεν θέλει να μετακινηθεί το Συμβούλιο. Ωραία, εγώ ακούω αυτά που λέτε, αλλά μπορούμε να του ζητήσουμε εμεί επίσημα να μετακινηθεί με ένα ψήφισμα, το οποίο θα ψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία και η οποία θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάει στο Συμβούλιο μετά και να το πει ορίστε. Πρέπει να μετακινηθείτε από τη θέση σα. Ε, το θέμα δεν είναι κανικότα το γοητευτικότα. Αν εμεί περιμένουμε το Συμβούλιο να μετακινηθεί που δεν μετακινείται, ε, προφανώ κινδυνεύουμε να ε, συνεχίσουμε πάπειρο την προσπάθεια και να περιμένουμε την επόμενη θητή και την επόμενη θητή και το καθεξής. Ας φροντίσουμε να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκείνο το οποίο... Εντάξει, δεν λέω ότι θα περάσει από μια κατάσταση όπου δεν έχει δικαίωμα σε ε, θέματα συνομοθέτη. Όχι, είναι συνομοθέτης, οπότε μπορεί κάλλιστα να πει αυτό θέλουμε. Το Συμβούλιο λυπάμαι, αλλά αδιαφορεί αν εμεί έχουμε αντιρρήσει τη μία μετά την άλλη και ενστάσεις όσο κερδίζει χρόνο. Ενώ εγώ, ναι, συμφωνώ, δεν είμαι σε θέση να αποφανθώ. Αλλά τι γίνεται, στο τέλος μιας διαδικασίας καταλήγουμε να εκφράζουμε αντίρρηση χωρίς να έχουμε παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία. Λοιπόν, για θέματα που δημοκρατικά είναι τόσο σοβαρά όσο είναι τα γενετικά τροποποιημένα που έχουν να κάνουν με την υγεία των ανθρώπων, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τη ζωή, ε, είναι πράγματα πολύ σοβαρά για να μην κάνουμε τίποτα. Δηλιάζει το Συμβούλιο. Ε, να του το πούμε και να απαιτήσουμε να κάνει κάτι. Και ο καλύτερος τρόπος είναι ένα ισχυρό ψήφισμα από τη δικιά μας την πλευρά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να θέλει το λόγο. Ε, Έγινε ανταλλαγή απόψεων, όπως προβλεπόταν σε μυρίσια διάταξη. Την είχαμε πράγματι αυτή την ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Οπότε βλέπουν τα πράγματα, βλέπουν οι, οι συνάδελφοι πώς έχουν τα πράγματα. Το σχέδιο έκθεσης θα το έχουμε το Φεβρουάριο στη συνεδρίασή μας. Εντάξει, είναι ξεκάθαρα αυτά. Ωραία, καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Και κάποια στιγμή στο μέλλον θα μάθουμε ποια θα είναι η συνέχεια. Ωραία. Τελειώνουμε έτσι με το σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη και περνάμε στο σημείο 6 που είναι η παρουσίαση από την Επιτροπή ε, σχετικά με την ευθύνη για την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες. Είναι εδώ, είναι εδώ. Ωραία. Η Επιτροπή μας παρακολουθεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ε, τεχνητή νοημοσύνη και τις άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες. Γι' αυτό και πολύ θέλουμε να ξέρουμε για την έκθεση της ε, νέας ε, ομάδας εργασίας για αυτά τα θέματα. Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει με έκθεση ιδίας νομοθετική πρωτοβουλίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε τον κύριο Τάρκ που είναι επικεφαλή τη Γενική Διεύθυνσης Just, που θα μας παρουσιάσει την έκθεση αυτή και μετά θα δώσουμε το λόγο στους ευρωβουλευτές για ερωτήσει και σχόλια. Παρακαλώ, αν είσαστε έτοιμο, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ε, με χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο μήνυμα και ακολουθούμε τώρα το ψήφισμα της Επιτροπής Τζούρι που θυμάμαι πάρα πολύ καλά το Φεβρουάριο του, 1900, 2017 όσον αφορά την πολιτική χρήση του ρομπότ. Και αν θυμάμαι καλά ήταν ένα ψήφισμα το οποίο έλαβε τεράστια προσοχή από το ευρύ κοινό και πραγματικά προσβλέπω στην ε, επικοδομητική συνεργασία που είχαμε τότε. Ε, να κάνω μία παρατήρηση. Το έγγραφο το οποίο μόλις σας μοιράσαμε, αυτή η έκθεση εδώ, δεν είναι, δεν είναι και πρέπει να το τονίσω αυτό, δεν είναι έγγραφο της Επιτροπής. Είναι η έκθεση μιας ε, ομα... ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει την Επιτροπή. Η Κομισιόν δεν έχει ακόμα ε, κάποια θέση, ε, εκτός από τις πολιτικές κατευθύνσεις που έδωσε η Πρόεδρος Βαντελάιεν. Αλλά για την ώρα δεν πρόκειται, επαναλαμβάνω, για έγγραφο της Επιτροπής. Αλλά με τα χαράς να σας εξηγήσω τι λέει αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων. Δύο λόγια σύντομα για το ποια είναι η πορεία. Η Κομισιόν υιοθέτησε τον Απρίλιο του 2018 μια ανακοίνωση για τις νέες ψηφιακές ε, τεχνολογίες, για τις πιθανές εργασίες μας περί αυτών, για την τεχνική, τεχνητή δηλαδή ευφυΐα, e e, είχαμε πρώτα τη βιομηχανική πολιτική, είχαμε μετά τις δεξιότητες και η τρίτη μας ανακοίνωση ήταν το κατάλληλο ηθικό και νομικό πλαίσιο, διοντολογικό μάλλον και νομικό πλαίσιο. Είχαμε ε, διοντολογικά και θεμελιώδη ε, δικαιώματα. Το, το, τρίτο το κομμάτι ήταν η ε, ευθύνη, ε, η οποία φυσικά συνδέεται με τα υπόλοιπα πολύ στενά. Χωρίσαμε σε δύο τμήματα την, έκθεση των ε, εμπειρογνωμόνων και αυτή η έκθεση είναι ε, η έκθεση εν... ενός από τα τμήματα, του δεύτερου τμήματο, πιθανές συστάσεις δηλαδή για τι, να κάνει η Επιτροπή με την ε, ευθύνη για την τεχνητή νοημοσύνη και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Πώς προχώρησε λοιπόν αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων. Καταρχάς, εξέτασαν τι ισχύουσε εθνικέ νομοθεσίε. Υπάρχουν διάφορε δικαιοδοσίε που εκπροσωπούνται στην ομάδα εμπειρογνωμόνων και μάλιστα είχαμε τη χαρά να έχουμε και παρατηρητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Επιτροπή Τζούρι. Και ε, όλοι εξέτασαν τι εθνικέ νομοθεσίε για να δουν και να αξιολογήσουν σε ποιο βαθμό οι ισχύουσε εθνικέ νομοθεσίε ε, μπορούν να ανταποκριθούν στι προκλήσει που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Σε μια δεύτερη φάση, προχώρησαν ε, για να εξετάσουν ε, ε, τις περιπτώσεις χρήσης ας πούμε τα αυτόνομα αυτοκίνητα, τα FEE, e, σπίτια, ιατρική έρευνα και ρομπότ, ντρόν κτλ δηλαδή πρακτικές εφαρμογές. Αφού είδαμε λοιπόν τις πρακτικές εφαρμογές και τις εθνικές νομοθεσίες ώστε να εντοπίσουμε τις προκλήσεις που δημιουργούνται λόγω της τεχνητής ευφυΐας, ε, νοημοσύνης, συζητήθηκαν διάφορες λύσεις και τα τελικά αποτελέσματα, όπως σας είπα, μόλις σας ε, διανεμήθηκαν. Εν συντομία να πω ότι η έκθεση και προσπαθώ να είμαι σύντομο ώστε να έχουμε χρόνο για ερωταπαντήσεις Να σας πω ότι καταρχάς λοιπόν η ομάδα πυρογνωμόνων ήρθε στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να επανεφευρεθεί ο τροχός. Οι νομοθεσίες έχουν ε, ασχοληθεί με τις νέες τεχνολογίες ανέκαθεν. Δεν χρειάζεται λοιπόν να δημιουργηθεί νέα βασική νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη, να ξεκινήσουμε από το μηδέν δηλαδή. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα στο οποίο έφτασε η ομάδα προγνωμόνων. Όμως ανέφερε επίσης η ομάδα προγνωμόνων διάφορες προκλήσεις που είναι ειδικέ και αφορούν ε, την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Μπορείτε να τα διαβάσετε αυτά στην έκθεση. Είναι διάφορες και πολλές και διάφορες. Οι προκλήσει είναι της αυτονομίας, της ε, αδιαφάνειας και της, του περίπλοκου χαρακτήρα. Αυτονομία τι σημαίνει? Ότι οι εφαρμογέ τεχνητή νοημοσύνης είναι σε θέση να λάβουν μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο να λάβουν αποφάσεις μόνε μόνες τους. Αδιαφάνεια σημαίνει ότι δεν είναι σαφές ούτε ακόμα και για αυτούς που τις φτιάχνουν πως μια τεχνητή νοημοσύνη, ένας αλγόριθμος φτάνει σε αυτή την απόφαση. Και αυτό είναι το εφέ του μαύρου κουτιού, όπως συχνά αναφέρεται στη συζήτηση. Και περίπλοκος χαρακτήρα σημαίνει ότι οι περισσότερες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται μέσα σε ένα περιβάλλον ίντερνετ των πραγμάτων. Ε, μπορεί να υπάρχουν δηλαδή υπηρεσίες και αγαθά και όλα αυτά μεταξύ τους συνδέονται. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να πάει πίσω και να δει τι έχει γίνει ακριβώς. Και αυτό είναι, εδώ σας τα απλοποιώ λίγο, αν θέλετε μπορείτε να μπείτε σε περισσότερες λεπτομέρειες στην έκθεση. Πάντως, συνδυασμένες αυτές οι τρεις προκλήσεις καθιστούν πάρα πολύ δύσκολη την ανακάλυψη, τον εντοπισμό ποιος, του ποιος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά συμβεί. Αυτό καθιστά επίσης πολύ δύσκολο το να ανοιχνεύσει κανείς στην αρχή που δηλαδή υπήρχε ένα ελάττωμα αν υπήρχε. Και ε, τέλος, επίσης πάρα πολύ δύσκολο για το θύμα να, να αποδείξει την αλληλουχία αιτίου αποτελέσματος μεταξύ ε, ενός ελαττώματος ενδεχόμενου ή μιας ζημιάς και, μάλλον, και της ζημιάς που τελικά έχει συμβεί. Οι προκλήσεις αυτές λοιπόν που έχουμε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το συνδυασμένο αποτέλεσμα, δηλαδή το συμπέρασμα της της ομάδας καταλήγει σε μια, ε, μια κατάσταση όπου είναι πιο δύσκολο αν όχι αδύνατον ή οικονομικός απαγορευτικό ένα θύμα να αποδείξει ότι είναι θύμα και να αποζημιωθεί για μια ζημιά η οποία έχει προκληθεί από μια εφαρμογή τεχνητής, νοημοσύνης. Και άρα λοιπόν σημαίνει ότι το θύμα δύσκολα ή σχεδόν ε, απίθανο είναι να έχει πραγματική πρόσβαση σε δικαιοσύνη και να δικαιωθεί. Βλέποντας λοιπόν όλες αυτές τις προκλήσεις, Λοιπόν, αν ε, λοιπόν Τώρα έχουμε ε, το δίκαιο περί που ισχύει ή ε, λέει ε, αν ας πούμε κάποιος, ε, κάποιον τον πατήσει αυτοκίνητο. Καταρχάς ε, πρέπει να δούμε τον οδηγό. Εάν ο οδηγός ε, ε, παραβίασε κάποιο φωτεινό σηματοδότη, τότε παραβίασε την νομοθεσία. Έπειτα έχουμε το αυτοκίνητο. Αν το αυτοκίνητο ήταν αλλοτοματικό και έπειτα ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Αυστηρή ευθύνη που υπάρχει σχεδόν και ισχύει σχεδόν σε όλα τα κρατημέλη ότι δηλαδή εδώ το θύμα δεν χρειάζεται να αποδείξει αν υπήρχε κάποιο σφάλμα ή κάποιο ελάττωμα, απλά μπορεί να διώξει ποινικά, το, ε, μάλλον να, να, καταγγείλει τον ιδιοκτήτη ε, του αυτοκινήτου για τη ζημιά που του προκλήθηκε. Τρεις διαφορετικές δυνατότητες υπό διαφορετικές προϋποθέσεις και εναντίον διαφορετικών δυνητικά υπεύθυνων ανθρώπων. Μόνο ένας εξ αυτών ε, είναι, ε, ένα εξ αυτών είναι εναρμονισμένο στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, την ευθύνη προϊόντος. Στα υπόλοιπα όχι. Και εκεί αυτή την περίπτωση εξέτασαν οι εμπειρογνώμονες και τι ε, τελικά που κατέληξαν. Είπαν ότι δεν χρειάζεται να επανεφευρεθεί ο τροχός. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε το δίκαιο περί αδικό πραξίας αλλά μπορούμε να τροποποιήσουμε τις ισχύουσε νομοθεσίες. Και προκύπτει λοιπόν ότι ε, προβαίνουν σε μια ενδιαφέρουσα διάκριση. Διάκριση σύμφωνα με το κίνδυνο των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Και άρα τις μοιράζουν σε αυτές που είναι υψηλού κινδύνου και αυτές που είναι χαμηλού κινδύνου. Και άρα ε, προτείνουν διαφορετικές τροπολογίες ανάλογα με το κίνδυνο που ενέχει η χρήση της κάθε εφαρμογή. δηλαδή μια προσέγγιση που βασίζεται στο κίνδυνο. Σας θυμίζω ότι αυτές είναι οι προτάσεις της ομάδας ε, των εμπειρογνωμόνων που ε, ασχολήθηκαν και με την δεοντολογία, δεοντολογία και την ε, νομοθεσία και εκείνοι βασίστηκαν σε μια τέτοια προσέγγιση κινδύνου. Ας δούμε λοιπόν, λένε πρώτα, τις εφαρμογέ υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, αυτές είναι μόνο κάποιες, δεν είναι όλες. Και ανέφεραν κάποια παραδείγματα όπου βασικά αυτές είναι οι εφαρμογές όπου εκτίθεται σε κίνδυνο περισσότερος ε, κόσμος και άρα όπου ε, διακυβεύονται σοβαρά πράγματα όπως η ζωή, η ασφάλεια, ή οικονομική ε, ζημιά σε ιδιοκτησία. Σε... Βασικά λοιπόν αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούν οι εμπειρογνώμονες ε, για να ορίσουν τις ε, εφαρμογές υψηλού κινδύνου. Μόνο λίγα παραδείγματα είναι οι εφαρμογές που κινούνται οι πιο επικίνδυνες. Δηλαδή τα αυτόνομα αυτοκίνητα, τα ντρόν, τα ρομπότ ε, παράδοσης πακέτων, δεμάτων και λίγα παραδείγματα. Τα περισσότερα, οι περισσότερες εφαρμογές είναι χαμηλού κινδύνου. Και εδώ απλοποιώ βέβαια γιατί τι εφαρμογέ υψηλού κινδύνου. Η ομάδα πυρογνωμονών προτείνει να επεκταθεί το μοντέλο που ισχύει αυτή τη στιγμή για τα παραδοσιακά αυτοκίνητα και σε αυτές τις εφαρμογές υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, αυστηρή ευθύνη για αυτές τις ε, ε, εφαρμογές υψηλού κινδύνου και ας το συνδέσουμε με την ασφάλιση προσώπων όπως γίνεται για τα παραδοσιακά αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα ότι το θύμα θα έπρεπε μόνο να αποδείξει ότι υπάρχει κίνδυνος στην... Ε, μάλλον ότι κάποιος από τους κινδύνους που προβλέπεται ότι μπορεί να ε, επιφέρουν αυτές οι ε, εφαρμογές υψηλού κινδύνου υπάρχουν και υλοποιήθηκαν, πραγματοποιήθηκαν. Και αυτό θα συνδέεται με υποχρεωτική ε, ασφάλιση. Δηλαδή η ιδέα θα ήταν ότι αν τώρα, ας πούμε, όπως τώρα, αν σε χτυπήσει αυτοκίνητο, η ασφάλιση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου είναι αυτή που σε αποζημιώνει. Και αυτό είναι ομαλό και πάει πολύ εύκολα. Ε, ε, και η ιδέα λοιπόν είναι να φτιάξουμε ένα παρόμοιο σύστημα. Αυτό, σε αυτό κατέληξε η ομάδα εμπειρογνωμόνων. Τώρα, για τις εφαρμογές χαμηλότερου κινδύνου, που είναι η μεγάλη μάζα. Ας πούμε, ε, ρομπότ ιατρικής έρευνας, εφή e σπίτια, αυτόνομες ε, μηχανές κουρέματος, γρασιδιού. Ας μείνουμε λοιπόν στο δίκαιο δικοπραξίας όπως ισχύει τώρα. λίγες προσαρμογούλες, ψηλοπροσαρμογούλες πρέπει να γίνουν ώστε να προσαρμοστεί το δίκαιο δικοπραξίας σε προκλήσεις ε, της ε, τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως αφορούν το πρόβλημα του βάρους της απόδειξης που αυτή τη στιγμή βαραίνει το θύμα. Οπότε βασικά υπήρξαν κάποιες εναλλακτικέ λύσεις και αρκετές εξ αυτών αφορούν, όπως είπα, το βάρος της απόδειξης. Βασικά λοιπόν προτείνουν διάφορες μεταβλητές για το πώς μπορεί να αντιστραφεί ή να ελαφρυνθεί το βάρος της απόδειξης. Μπορεί να είναι γενικευμένο το βάρος της απόδειξης, μπορεί να μετακινηθεί το βάρος της απόδειξης. Η ελάφρυνση όπως σας είπα σε συγκεκριμένες υποθ... περιπτώσεις. Και είναι η εξής. Για παράδειγμα, είναι ενδιαφέρον το συνδέουν με μια υποχρέωση εισόδου, το logging. Ήδη ε, το έχουν προβλέψει κάποιοι παραγωγοί όταν ας πούμε υπάρχουν ε, ημέρες δοκιμής, ας πούμε, ε, για τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Λέει λοιπόν 15 λεπτά πριν το ατύχημα. Η ιδέα είναι να πούμε ότι εφόσον έχεις βάλει αυτά τα στοιχεία, τα δίνεις τα δεδομένα στο θύμα, ώστε το θύμα να μπορεί να αποδείξει την υπόθεση του. Αν όμως δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα ή αν δεν θέλεις να τα δώσεις στο, στο, θύμα, τότε αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης. Η άλλη ιδέα είναι να συνδεθεί με την κυβερνοασφάλεια ή την ασφάλεια των προϊόντων που θα χρειαστεί να προσαρμοστεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά οι κανόνες ε, κυβερνοασφάλειας που θα προσαρμοστούν και ας πούμε θα προσαρμοστούν με το γεγονός ότι τα προϊόντα ε, εξελίσσονται. Υπάρχουν διαρκείς ε, ενημερώσεις, updates Παίρνει λοιπόν ένας από, ένα θύμα, ε, ειδοποιήσει ότι πρέπει να κάνει update και δεν το κάνει. Εκεί σημαίνει ότι παραβιάζει τα στάνταρ κυβερνοασφάλειας, πράγμα το οποίο βαραίνει τον ε, ε, χειριστή, το φορέα διαχείρισης. Εφόσον τα έχει κάνει αυτά όπως πρέπει όμως ο φορέας διαχείρισης, εντάξει, το έχει κάνει, αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα, άρα το θύμα θα πρέπει να αποδείξει. Αν όμως ο φορέας διαχείρισης δεν έχει κάνει την ενημέρωση, δεν συμμορφώνεται προς τις κανόνες ασφάλειας, τότε αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης. Ε, κάποια, απλώς αυτά είναι κάποια παραδείγματα και προτάσεις όπως σας είπα. Να σας αναφέρω τέλος κι άλλο ένα παράδειγμα. Ότι αυτό που αφορά την ε, ευθύνη ε, όπως ας πούμε για ένα ρομπότ ε, για ε, εγχειρήσεις. Αν είσαι γιατρός, ένας γιατρός άνθρωπος κάνει λάθος, μπορεί κανείς να διώξει τον γιατρό αλλά και το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι υπεύθυνο διότι ο γιατρός είναι ο υπάλληλό του. Και σε πάρα πολλές χώρες υπάρχουν βέβαια διαφορετικοί κανόνες που όμως τελικά καθιστούν τον εργοδότη υπεύθυνο για το τι κάνει ο εργαζόμενός του, για λάθος του εργαζόμενου του. Οι υπερογνώμονες λένε όμως αυτό δεν θέλουμε να το αγγίξουμε. Αυτό θα πρέπει να μείνει η εθνική νομοθεσία ω έχει. Οι κανόνες διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Α τα αφήσουμε έτσι. Όμω, αν το νοσοκομείο αντικαταστήσει τον άνθρωπο γιατρό από εφαρμογή τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα πρέπει να ξεφύγει από τις ευθύνες του απλά και μόνο επειδή αντικατέστασε τον άνθρωπο από μηχάνημα. Αυτό το λέμε ε, ε, human equivalence, ανθρώπινη αντιστοιχεία. Ε, αντιστοιχεία της ευθύνης. Είναι μια από τις πολλές προτάσεις τις οποίες κατέληξε η ομάδα των εμπειρογνωμών. Όπως είπα και πριν, τονίζω και πάλι ότι δεν είναι έγγραφο της Κομισιόν. Είναι έγγραφο μιας ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμών που συμβουλεύει την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στάτομα για πάρα πολύ ε, χρήσιμη ε, και διαφωτιστική παρέμβασή σας να ξεκινήσουμε. Μελχιόρ, μιλήσατε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ε, σε χειρουργικές επεμβάσεις ε, στο τέλος. και όταν μιλήσατε για κάποιες υψηλού κινδύνου εφαρμογές, έχω μια ερώτηση. Αν χρησιμοποιούνται σε συνεργασία με ιατρικές εφαρμογές που δεν κινούνται όπως ίσως τα αυτόνομα αυτοκίνητα, όμως υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και τη ζωή του ανθρώπου αν κάτι δεν πάει καλά. Άρα με τη σύσταση θα υπάρχει αυτή η αρχή της οτιμίας, της ισοδυναμίας ή θα πρέπει ε, να χρησιμοποιηθεί για τη, το τεχνολογικό εξοπλισμό και τις σχετικές εφαρμογές ε, το δίκαιο περιοδικό πραξιών. Και υπάρχει αυτό το μαύρο κουτί όταν μιλάμε ε, για την τεχνητή νοημοσύνη που έχει να κάνει με μηχανήματα. τι σκέφτεστε όταν χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη. Ε, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τι κάνει. Δηλαδή, μια τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξηγεί τι κάνουν οι άλλες συσκευές τεχνητής νοημοσύνης. Και ένα θέμα που θέλω να θίξω, που αφορά τη Δανία πιο πολύ, που έχουμε δυνατότητα εξαίρεσης ό,τι αφορά τη συνεργασία στο τομέα του αστικού δικαίου. Υπάρχουν προτάσεις νέας ε, νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να εμπίπτουν σε, αυτή, το, σε αυτό το δικαίωμα εξαίρεσης της Δανίας, άρα να μην ισχύσουν στην περίπτωση της χώρας μας. Απάντησα. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Καταρχάς, η ομάδα εμπειρογνωμόνων όταν μελετά για ε, την ευθύνη κοιτάζει κυρίως τις ε, εφαρμογές υψηλού κινδύνου και εκεί συνδυάζει στοιχεία τα οποία είναι πρώτα απ' όλα η έκθεση του πλατιού κοινού στον κίνδυνο και δεύτερον αν ε, είναι υψηλού συμφέροντος ε, και αξίας ε, αυτό το οποίο τίθεται σε κίνδυνο, η ζωή, η υγεία ή κάποιο πολύ σημαντικό αγαθό. Και τώρα υπάρχει το σωρευτικό αποτέλεσμα, παρότι αυτό δεν λέγεται ξεκάθαρα, που σημαίνει ότι η άμεση αυτή αυστηρή ευθύνη στην έκθεση της Επιτροπής Επιγραμμών ισχύει για σωρευτική συνδυασμό αυτών των δύο στοιχείων. Στο δικό σας παράδειγμα δηλαδή, ε, όταν έχουμε τα ρομπότ που κάνουν ε, χειρουργική επέμβαση, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο νόμο συμφέρον, υγεία, ζωή, αλλά δεν κινδυνεύει το πλατή κοινό, το ευρύ κοινό. Αλλά ο συγκεκριμένος, μεμονωμένος ασθενής. Εδώ λοιπόν, νομίζω το συμπέρασμα της ε, ομάδας των είναι ότι είναι χαμηλής ε, επικινδυνότητας, όχι ότι δεν είναι σημαντικό, ε, είναι ταξινόμηση ουσιαστικά. Το δίκαιο περί αδικοπραξιών εδώ ισχύει, αλλά με μικρές στοχευμένες προσαρμογές, αυτές που σας ανέφερα. Δεύτερον, για το μαύρο κουτί και την ε, εκμάθηση, το machine learning από τις μηχανές. Καλό και σημαντικό είναι να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ, και γι' αυτό είπα ότι ένας από τους πολλούς λόγους ε, που είπα τέλο πάντων ότι είναι πολύ στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους οι διάφορες ε, διαστάσεις του θέματος και πρέπει να προχωρήσουμε με βάση όλες αυτές τις διαστάσεις. Εδώ μπορώ να σας αναφέρω το έργο της ομάδας ψηλού επίπεδου που συγκρότησε η Κομισιόν με ένα σημαντικό σκέλος ακριβώς ε, αυτό που αναφέρατε, δηλαδή το να μπορούμε να παρακολουθούμε να ελέγχουμε, να εξηγούμε κατά βάση πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική πτυχή σε ό,τι αφορά το δανέζικο opt-out. Δεν είμαι ειδικό, αν θυμάμαι καλά όμως, αφορά τη δικαστική συνεργασία, τον εν λόγω τίτλο, και όχι νομικές πράξεις που βασίζονται στο 114 άρθρο της συνθήκης. Βέβαια, αυτό που σας παρουσιάσαμε, παραλαμβάνω, είναι μια έκθεση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων. Δεν είναι επίσημη γραμμή της Κομισιόν. Δεν μπορούμε να πούμε τι ε, πιστεύει για αυτή την πρόταση η Κομισιόν. Και αυτή και είναι και η απάντηση που μπορώ να σας δώσω. Και το μόνο που θυμάμαι είναι ότι υπήρχε ένα ψήφισμα της Επιτροπής Γιούρη το Φεβρουάριο του 2017 που ζητούσε να καταθέσει η Κομισιόν πρόταση δυνάμει του άρθρου 114, αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Δεν υπάρχει γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνητή νομοσύνη, το λέω ξεκάθαρα. Θα υπάρξει τοποθέτηση εκ μέρους Κομισιόν, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο τις πολιτικές κατευθύνσεις της Προέδρου, που πράγματι ανακοινώνει συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για τι ανθρώπινε και τι ειδικέ πτυχέ ε, τη τεχνητή νοημοσύνη. Ευχαριστώ. Κάρεν, μήπω θέλει να επανέλθει, Αν όχι, ε, έχουμε και άλλους ε, γι' αυτό. Καλό θα ήταν να μην ξαναπαρσταλώ. Ναι, εγώ, λέει η κυρία Βάλσμαν, και αφού ευχαριστήσω τον κύριο Στατμάιερ για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Ε, θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα τα οποία μου προκάλεσαν ενδιαφέρον. Πρώτον το θέμα της κυβερνοασφάλειας που για μένα είναι κάτι ουσιώδες και όταν μιλάμε για το ε, διαδίκτυο των πραγμάτων, το ίντερνετ των πραγμάτων δεν έχουμε μόνο τη σχέση μεταξύ κατασκευαστή και χρήστη, αλλά έχουμε και ένα ρομπότ που δίνει ε, μέσω καθοδήγησης ε, ε, μια εντολή σε ένα άλλο ρομπότ για να κάνει κάτι. Δηλαδή έχουμε δύο μηχανήματα, δύο συσκευές, δύο ρομπότ που επικοινωνούν. Και έχουμε και το θέμα της ασφάλειας δεδομένων που γίνεται πολύ λόγος. Ε, όχι στον αρχικό προγραμματισμό μόνο, αλλά και στην εκμάθηση και αν υπάρξει ε, κάποιο είτε ε, δεδομένο σκόπιμο, είτε ένα σφάλμα τέλο πάντων, και αν ε, υπάρχει και ένας τρίτος που εμπλέκεται δεν είναι εύκολο να ε, αποδοθεί ευθύνη. Και όταν έχουμε λοιπόν ε, την καθοδήγηση, έξωθεν καθοδήγηση, εντολή ενός ρομπότ, ποιος έχει την ευθύνη. Και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση της επικινδυνότητας. Μιλήσατε ε, για τις ε, χορτοκοπτικές μηχανές που τις κατατάξατε στις χαμηλού κινδύνου εφαρμογές. Θα μπορούσε ένα ρομπότ να είναι ε, μια ασφαλής εφαρμογή, αλλά αν έχουμε παιδιά που παίζουν ή κατοικίδια που μπορεί να είναι θύματα, να υποστούν κάποια βλάβη, τελικά ε, δεν ξέρω κατά πόσον είναι επαρκής αυτή η κατηγοριοποίηση να μιλάμε ίσως μόνο για ε, τη χρήση ή το χρόνο. Θα πρέπει να δούμε και την ταξινόμηση επίσης. Ποιος αποφασίζει τι είναι ασφαλές μηχάνημα, ποια είναι ασφαλή συσκευή. Ε, να, τέτοιο χορτοκοπτικό μηχάνημα που ε, μπορεί να έχει και επαφή με τον νερό κτλ. Δεν ξέρω, ε, μπορεί να υπερβάλλω, απλά θέλω να σας το καταστήσω σαφές ότι ε, αυτό για μένα είναι ένα αποφασιστικό σημείο. Ποιο είναι αυτό ο οποίο αναλάβει την ευθύνη για αυτήν την ταξινόμηση και αυτό που την αναλαμβάνει δεν νομίζω ότι έχει και την αστική ευθύνη τελικά. Ευχαριστώ πολύ τι ερωτήσει σα. Καταρχά, σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια και το διαδίκτυο των πραγμάτων, αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας και πάρα πολύ ε, σωστά είπατε ότι μεταξύ πολλών άλλων προβλημάτων υπάρχει εδώ και το πρόβλημα το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς ε, ε ποιος έχει κάνει κάτι. Και αν το βρει υπάρχει μια πρόσθετη δυσκολία να υπάρχει και ένας hacker, για παράδειγμα, που έκανε κάτι, που ούτε μπορεί να τον βρει κανείς ή δεν μπορεί να πληρώσει. Ε, είναι αφαιρέγγιος. Ε, και αυτό ε, το αναφέρουν στην εκθεσή τους οι εμπειρογνώμονες και αναφέρουν κάποιες δυνατότητες έτσι πολύ διερευνητικά για το τι θα μπορούσε να γίνει Ähm, Στην περίπτωση που δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ο hacker ή δεν μπορεί να ε, πληρώσει, ε, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει ε, κάποια άλλη λύση, με οτιδήποτε. Αλλά αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες ότι αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αυτό το οποίο θίξατε και πραγματικά πολύ προσεκτική και διατύπωση στο κείμενο αυτής της έκθεσης για το θέμα αυτό. Επίσης μιλήσατε για τη συμμετοχή τρίτων, αν δεν είναι δηλαδή το σφάλμα στον αρχικό προγραμματισμό. Πράγματι ισχύει αυτό ε, και έχουμε και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Ε, δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα μπορεί να υπάρξουν σφάλματα. η τεχνητή είναι λειτουργεί όπως θα έπρεπε ε, και δεν υπάρχει εδώ κάποιο σφάλμα. Υπάρχουν κάποια ε, προσπάθειες να ε, χρησιμοποιηθούν ρομπότ ε, για την καθαριότητα των δρόμων του Δήμου. Αν πούμε ότι είναι ένα στενός δρόμος και βγαίνει και τρέχει στο δρόμο ένα παιδάκι, το ρομπότ έχει έναν αλγόριθμο που είναι έτσι σχεδιασμένος που του ε, λέει ότι πρέπει να αποφύγει, παρακάμπτει το, το παιδί, δεν μπορεί να κάνει κακό ε, αλλά αν ας πούμε προκύψει ε, βλάβη ε, σε ένα όχημα, τι γίνεται. Αν έχει λειτουργήσει όμως ε, το μηχάνημα αυτό, η τεχνητή νομοσύνη όπως έπρεπε, αλλά δημιουργηθεί παρόλα αυτά βλάβη, ζημία, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Όταν είναι ένα πρόβλημα. Και όταν επίσης έχουμε πολλούς οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα πολύπλοκο οικοσύστημα όπως είναι το ίντερνετ των πραγμάτων, τότε πράγματι υπάρχει το ερώτημα και όχι μόνο για τους hacker. Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε, να ταυτοποιήσουμε τον υπεύθυνο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό και πρέπει να κινούμαστε πολύ προσεκτικά σε αυτό το έδαφος και σε ό,τι αφορά τα χορτοκοπητικά, των μηχανές κουρέματος και ποιος είναι ο, ε, αυτός που έχει την αστική ευθύνη. Ναι, πράγματι. Όταν έχουμε αυτόνομα, τέτοιε μηχανές μπορεί να προκύψουν ατυχήματα. Και νομίζω υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα ε, στον τύπο ότι δοκιμάστηκαν 10 τέτοια ε, μηχανήματα σε ένα πλαστικό μωρό, κούκλα, που ήταν στο γρασίδι ε, και σε δύο περιπτώσεις πάτησε τα πλαστικά πόδια η μηχανή. Υπάρχει δηλαδή και αυτό το ενδεχόμενο. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αυτό το σφάλμα δεν το κατέταξε στα υψηλού κινδύνου γιατί δεν πλήττεται το πλατή κοινό, όπως είπα. Αλλά αυτοί οι οποίοι κορεύουν το γρασίδι, προκεκλημένοι ενδεχομένω του ιδιοκτήτη. Άρα ε, το δίκαιο περιαδικοπραξίας εδώ θεωρείται επαρκές, με μικρές προσαρμογές από την ομάδα εμπειρών, που κάνει την ταξινόμηση. Χμα. Καταρχήν, αυτό μπορώ να σας πω και πόσες φορές θα το επαναλάβω, είναι ότι αυτή είναι απλά μια έκθεση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων. Και σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε ότι αυτό πρέπει ε, να ε, γίνει ε, ένας κανόνας που θα επιβληθεί. Ότι αυτή είναι μια καθοδήγηση. Αλλά σίγουρα η ταξινόμηση είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Και αν ε, γίνει ε, κάτι λάθος. Ε, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολιτική κατά βάση αυτή. Σας ευχαριστώ. Thank you. Um, Mr. Voss is next. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριος Voss. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχηθώ και σας, κύριε Στατμάιερ, καλή χρονιά. πολύ καλή επιλογή για αυτό το θέμα στην αρχή της νομοθετικής της θητείας που το εξετάζουμε το θέμα αυτό της ευθύνης. Δεν ξέρω κατά πόσον το ίδιο προκύπτει και την έκθεση, αλλά δική μου άποψη είναι. Και αν η ομάδα εμπειρογνωμών παραπέμπει σε διάφορες λύσεις ή ε, κανόνες ε, που μπορεί να ισχύουν στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την αστική ευθύνη. δεν ξέρω κατά πόσο είναι επαρκή αυτό επιχείρημα. Όταν έχουμε την εποχή της παγκοσμιοποίησης και όταν έχουμε εφαρμογές ε, και ε, μεταφορά δεδομένων χωρίς κανένα όριο ε, ότι θα ε, έχουμε έναν κατακαιρματισμό ε, στο πλαίσιο της αγοράς. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό. Το έχουμε ξαναζήσει και στην προηγούμενη θητεία και δεν θέλουμε να το επαναλάβουμε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή να έχουμε κάποιες οδηγίες, αλλά όχι. Πρέπει να το δούμε σοβαρά αυτό το θέμα στο πλαίσιο της αγοράς και να προσπαθήσουμε να βρούμε αρμονισμένους ενιαίους κανόνες Δεν θέλει η ομάδα μου να περιοριζόμαστε σε οδηγίες, αλλά να προχωρήσουμε ε, σοβαρά ε, στην ανασχόλησή μας ε, με τους κανόνες εσωτερικής αγοράς. Όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, σίγουρα εδώ οι διατάξει εφαρμόζονται θεσνοριακά. Και δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός. Ποιος ευθύνεται, γιατί, τι καθεστώς ευθύνης ισχύει, θα χάσουμε τον μπούσουλα. Ε, επομένως, ε, κανονικά θα έπρεπε να στοχεύουμε στην εναρμόνιση και... Έρχομαι και σε ένα άλλο ερώτημα, αυτό της Μάριαν Βάλτσμαν, με την ταξινόμηση της επικινδυνότητας. Είναι αναγκαίο να υπάρχει μια τέτοια πολυπλοκότητα σε αυτόν τον κανονισμό, που τελικά κανένας δεν ξέρει τι δικαιώματα έχει, πού τα έχει, σε ποια χώρα και ε, αν ε, είναι υψηλή, ή χαμηλής επικινδυνότητας ε, κτλ. κτλ. Δεν βοηθάει αυτό. Δεν θα πρέπει την νομική δομή να την περιπλέκουμε στο διηνικές με αυτόν τον τρόπο, αλλά πρέπει να στοχεύσουμε αντίθετα σε πιο απλές λύσεις. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση που μπορεί να δικαιολογείται, αλλά αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε να απλωστεύσουμε αντί να διαφοροποιούμε ε, και να προσπαθούμε εθνικά να ε, ρυθμίσουμε το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά επίσης το ψηφιακό περιεχόμενο, μιλήσαμε για τις ενημερώσεις και στην προηγούμενη θητεία. Αν κάνουμε αυτή τη σύγκριση και λέμε έτσι είναι τα πράγματα για τα οχήματα, υπάρχουν κάποια συστήματα αστικής ευθύνης κτλ. αλλά ε, αν τα φρένα δεν λειτουργούν ε, καλά πρέπει να πάω στον ε, κατασκευαστή για να τα βελτιώσει λοιπά. Υπάρχει πρόβλημα ενδεχομένως με κάποια ζητήματα, με κάποιους μηχανισμούς ή συστήματα και χρειάζεται μια ενημέρωση, ένα update, αλλά τελικά το βάρος ποιος το φέρει και πρέπει να πληρώσει. Τι γίνεται στην περίπτωση τεχνητή νοημοσύνης. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις ή να προχωρήσουμε σε μια απλούστευση για να ξέρει ο πάσα ένας τελικά ε, τι δικαιώματα έχει και τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Και με αυτό το login που μας ε, παρουσιάσατε, δηλαδή ουσιαστικά η ομάδα εμπειρογνωμών παρουσιάζει, Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει ε, υποχρέωση, υποχρεωτική καταχώρηση ε, και πρωτοκόλληση. να υπάρχει αυτό, ε, αυτή η καταγραφή υποχρεωτική. Το σημαντικό για μένα όμως είναι να έχουμε κανόνες νέους για την εσωτερική αγορά. Να μην μιλάμε μόνο γι' αυτό, ούτε να έχουμε αυτά τα 27 διαφορετικά συστήματα. να είναι πολύ τα πράγματα μόνο εκεί που δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Αλλιώ να προχωρήσουμε με πιο απλέ λύσει. Αρκά, αρκετά περίπλοκο είναι ο κόσμο όπω έχει. Thank you. very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Να σας ε, αντευχηθώ κι εγώ, κύριε Φως. Το πρώτο ερώτημα είναι πολιτικού χαρακτήρα και δυστυχώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ επ' αυτού. Ε, γνωρίζουμε όμως από τις ε, συνομιλίες μας στα κρατημέλη ότι γίνεται και στα κρατημέλη συζήτηση για το κατά πόσο είναι προσαρμοσμένα αυτά τα συστήματα αστικής ευθύνης ε, στις απαιτήσει της τεχνητής νομοσύνης. Άρα γίνεται αυτή η συζήτηση. Δεύτερο θέμα για την ταξινόμηση. Ε, πολύπλοκοι κανόνες λέτε. Ναι. Μα είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα. Τι να κάνουμε. πώς θα λύσουμε το γόρδιο δεσμό εδώ, ε, πώς θα βρούμε ε, μια απλή λύση ε, αντικειμενική. Εγώ θέλω να σας επιστήσω την προσοχή σας σε μία πρόταση της Ομάδας Συμπρογραμμόνων για την νοημοσύνη, δηλαδή την διατήρηση της ισορροπίας αφενός μεταξύ μίας δίκαιης αποζημίωσης για τα θύματα ε, δηλαδή να αποζημιώνεται δίκαια αντίστοιχα με την αποζημίωση που θα έπαιρνε ε, αν είχε υποστεί βλάβη ε, από ένα παραδοσιακό μέσω της παραδοσιακού σε εφαρμογή ή τρόπου. Και το θέμα είναι, έχουμε και την ανακοίνωση του 18 για τεχνητή νοημοσύνη όπου λέει η Κομισιόν ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε το δυναμικό της τεχνητής νομοσύνης. Άρα, όταν ε, είναι δυνατόν, θέλουμε να προτείνουμε και πολιτικά μέτρα τα οποία θα προωθούν την καινοτομία. Αυτή είναι οι δύο βασικοί πολιτικοί στόχοι που πρέπει να είναι ισορροπημένοι μεταξύ τους. Γι' αυτό τότε υπήρχε και αυτή η ομάδα υψηλού επίπεδου για την τεχνητή νομοσύνη, η οποία είχε προτείνει για όλες τις ιδέες, προτάσεις στον τομέα αυτό, να υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση επικινδυνότητας. Και γι' αυτό έχουμε high risk, low risk, υψηλή χαμηλή επικινδυνότητα και αυτή την ταξινόμηση. Αλλά είναι πολιτικό το θέμα και εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο από αυτού. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ενημερώσεις ε, και τα updates και τις υποχρεώσεις. Πράγματι, έχουμε τις ε, οδηγίες για το ψυχικό περιεχόμενο και για τα εμπορεύματα με ψηφιακό περιεχόμενο. Πράγματι ε, υπάρχει αυτή η υποχρέωση για ε, ενημερώσεις και εκεί, αν θυμάστε, προβλέπεται και αυτή η αποζημίωση ότι αρχικά ο έμπορος είναι αυτός ο οποίος υποχρεούται να ε, ετοιμάζει και να διαθέτει τις ενημερώσεις. Σίγουρα αυτό είναι ένα άχθος, είναι ένας φόρτος εργασίας, γιατί συνήθως αυτό κάνει ένας τρίτος, δεν το κάνει ο ίδιος ο ε, εμπόρος και απ' την άλλη ο όταν δεν εγκαθιστά αυτές οι ενημερώσεις μπορεί να ε, ζητήσει αποζημίωση ή να προσφύγει και να ζητήσει ε, την αποζημίωση αν υπάρξει πρόβλημα. Αυτή είναι η απόφαση του νομοθέτη. Η ενημερώση σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα και για την τεχνητή νομοσύνη, αλλά και για άλλε αναδυόμενε τεχνολογίε. Διότι τα προϊόντα στη διάρκεια του κύκλου ζωή του με τι ενημερώσει βελτιώνονται. Ε, είτε ε, από τους ε, φορείς, είτε από τους καταναλωτές, είτε από τους κατασκευαστές, είτε από οποιοδήποτε τρίτο υπάρχουν αυτές οι ενημερώσεις διαθέσιμες και σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα να δούμε τι κάνουμε, αλλά υπάρχει στις οδηγίες μία πρόταση για την αποζημίωση σε περίπτωση προβλήματος. Και το τελευταίο για αυτή την ε, ταξινόμηση ή το πρωτοκόλληση, τέλο πάντων την καταγραφή, αυτό το login, αυτή την υποχρέωση. Πάντα λαμβάνοντα υπόψη τι διατάξει του Γενικού Κανονισμού Προστασία Δεδομένων. Θα πρέπει να αποθηκεύονται κάποια δεδομένα τα οποία πρέπει να δοθούν στο θύμα. Και αν αυτό δεν γίνεται, τότε υπάρχει αυτή η μετατόπιση, είπαμε, η ελάφρυνση του βάρου απόδειξη. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν ε, εδώ για ένα τόσο σημαντικό θέμα, λέει ο κύριος Διδιέ. Αναφερθήκατε στη δυνατότητα ανατροπής του βάρους της απόδειξης σε κάποιες περιπτώσεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτός που έχει το βάρος της απόδειξης πρέπει να αποδείξει αυτό που υποστηρίζει και όχι ο άλλος να αποδείξει την ε, αθότητά του. Καταλαβαίνω ότι πάντα υπάρχουν ε, εξαιρέσεις σε παντός είδους δίκαιο, αλλά το ερώτημά μου εδώ είναι το εξής. Εσείς έχετε καθορίσει κριτήριο επί της αρχής που σας ε, επιτρέπει να υποστηρίξετε ότι όταν υπάρξουν εξαιρέσει θα είναι κατά περίπτωση, θα είναι ανάλογα με την οικονομική επιβάρυνση της ευθύνης ή βάση κάποιων άλλων κανόνων. Γιατί εγώ για άλλη μια φορά πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι κατά του να υπάρχουν εξαιρέσεις όσον αφορά αυτό το βάρος της απόδειξης. Είμαι όμως πεπισμένος ότι οι εξαιρέσεις αυτές άπαξ και υπάρχουν θα πρέπει να πλαισιώνονται δεόντως. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας ε, αυτή. Αναφέρατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πράγματι, την αρχή του βάρους της απόδειξης που επιβάλλεται σε αυτόν που ζητάει. Ε, στο θέμα λοιπόν αυτό είναι τα θύματα που ε, πρέπει να καθορίσουν τα διάφορα κριτήρια για να καθοριστεί το θέμα της ευθύνης. Όμως υπογραμμίσατε συγχρόνως και πολύ σωστά ότι πράγματι έχουν ήδη προβλεφθεί εξαιρέσεις Στη Γαλλία, για παράδειγμα, στο θέμα της εξωσυμβατικότητας στον ιατρικό κόσμο, αλλά και αλλού. Πολλές φορές υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις και ο Μάτι Περογνωμόνων συζήτησε πολύ σε βάθος αυτά τα ζητήματα, όπου ακριβώς εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της κατάστασης, το θύμα αντιμετωπίζει δυσκολίες ανυπέρβλητες ή περίπου προκειμένου να αποδείξει ότι έχει δίκιο. Και το εθνικό δίκαιο ε, πράγματι προβλέπει εξαιρέσεις παντός είδους και φύσεως και ακριβώς γι' αυτό η ομάδα πυρογνωμόνων δεσμεύτηκε προς αυτή την κατεύθυνση της συζήτησης, γιατί είδαν ότι υπάρχουν προηγούμενα που υπάρχουν ήδη στα διάφορα εθνικά δίκαια. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερον, με ρωτάτε αν καθορίσαμε κριτήριο. Αν είσαστε εσείς η Επιτροπή, και επιμένω που το λέω και το ξαναλέω αυτό, επιμένω ότι εμείς τίποτα δεν καθαρίσαμε. Γιατί δεν έχουμε αποφασίσει τίποτα από αυτού. Πρόκειται για την ομάδα εργασίας, η οποία πρότεινε κάποιες ιδέες πάνω στις οποίες να προβληματιστούμε. Αλλά είναι σαφές ότι αν προχωρήσουμε σε αυτόν τον προβληματισμό, που θα είναι είτε συσσωρευτικά είτε εναλλακτικά, σίγουρα πρέπει να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και να δούμε πώς ε, μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά με περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτά προς το παρόν. Υπάρχουν ιδέες για προβληματισμό που πρότεινε η ομάδα εμπειρογνωμόνων. Αναφερθήκατε εσείς σε κριτήρια, σε δυνατότητες ή σε καταπερίπτωση, ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης ή αν θα υπάρχουν κάποια κριτήρια επί της αρχής. Εγώ δεν έχω άποψη από αυτού, αλλά είναι σαφές από τις συζητήσεις που έγιναν στην ομάδα περιγνωμόνων ότι η νομική ασφάλεια για την ομάδα αυτή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέλημα. Πράγματι, συζήτησαν μήπως θα μπορούσαν να τα αφήσουν στην εθνική ε, δικαιοδοσία που θα αποφάσισε κατά περίπτωση. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, αλλά είπαν επίσης στη συζήτηση ότι υπάρχει ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση να μην δημιουργηθεί νομική ασφάλεια. Δηλαδή, εντάξει, θα υπάρχει κάποια λύση νομική κατά περίπτωση, αλλά δεν θα υπάρχει νομική ασφάλεια. Είμαστε εδώ σε μία, πώς να το πω, σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν δύο σημαντικές αρχές που με κάποιο τρόπο πρέπει να συνεπάρξουν. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο από αυτόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λεμπρετό και μετά ο κύριος Γκονζάλης Πόνς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, είναι σημαντικό να σκεφτούμε αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως όπως κάνουμε και σήμερα, να δούμε τι γίνεται με την αστική ευθύνη εφόσον υπάρξουν βλάβες από τα αυτόνομα ρομπότ. Εγώ εδώ συγκράτησα διάφορες ιδέες που προτείνει η έκθεση εμπειρογνωμόνων. Κυρίως την ιδέα να υπάρχει μια υποχρεωτική ασφάλιση ή επίσης μια άλλη ιδέα πρέπει να σκεφτούμε να υπάρξει και αντιστροφή του βάρους της απόδειξης υπέρ των θυμάτων. Ωραία. Όμως εγώ έχω και άλλες ερωτήσεις. Δύο κυρίως. Η πρώτη μου. Όταν είχαμε προβληματιστεί για αυτό το θέμα της ε, αστικής ευθύνης στην προηγούμενη θητεία, κάποια στιγμή σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε ενδεχομένω να υπάρχει ε, μία νομική προσωπικότητα για τα ρομπότ. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν συμφωνίες, ξέρω για μία ανοιχτή επιστολή στην Επιτροπή από 300 ερευνητές για την τεχνητή ε, νοημοσύνη ε, που δήλωναν κατά μια τέτοια ιδέα. Πού βρίσκεται ο προβληματισμός από αυτού. Δεύτερον, πιο συνολικά έχουμε ήδη μία οδηγία που υπάρχει και είναι εκείνη που αφορά τα λατωματικά προϊόντα και που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των ε, ρομπότ. Ποιος όμως αξιολογεί τελικά αυτή την οδηγία. Είναι εξωτερική υπεύθυνη και μήπως εδώ πέρα τίθεται θέμα αντικειμενικότητας. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ε, ερώτησή σας. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων όντως γνωρίζει την επιστολή αυτή των ερευνητών στην οποία αναφερθήκατε εσείς. Και έγινε συζήτηση επ' αυτής. Και μπορώ μάλιστα να σας πω ότι, γιατί εδώ ναι έχω μια θέση από πλευρά Επιτροπής, γιατί αντιδρώντας το ψήφισμά σας του Φεβρουαρίου του 2017 που ήδη ανέφερε το θέμα της νομικής προσωπικότητας, ήταν πολύ διστακτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων λοιπόν πήγε προς την ίδια κατεύθυνση και μάλιστα ακόμα πιο έντονα. Δεν πιστεύει δηλαδή ότι μια τέτοια νομική προσωπικότητα για τα ρομπότ είναι κάτι που όντω είναι κατάλληλο για το θέμα που συζητάμε. Το κύριο επιχείρημά του στη συζήτηση ήταν ότι σε τι θα βοηθήσει. Γιατί αν δημιουργήσουμε μία νομική προσωπικότητα, απλώς αναβάλουμε το πρόβλημα. Γιατί αν δημιουργήσουμε μια τέτοια νομική προσωπικότητα, θα πρέπει αυτή η νέα προσωπικότητα να συνοδεύεται και από κάποια κονδύλια, ώστε να μπορεί να υπάρξει αποζημίωση της λάβης. Ποιος θα πληρώσει. Οπότε και πάλι πρέπει να βρούμε κάποιον που θα πληρώσει. Ε, και τότε ποιο θα είναι, θα είναι ο υπεύθυνο. Οπότε γιατί να δημιουργηθεί και αυτή η νομική προσωπικότητα επιπλέον. Πάντω, σαφώ η ομάδα πυρογνωμόνων είναι κατά τη ιδέα αυτή για νομική προσωπικότητα ε, στα ρομπότ. Τώρα έρχομαι στο θέμα της αξιολόγησης της οδηγίας για τα ελαττωματικά προϊόντα. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει ε, μια έκθεση για την αξιολόγηση της ε, οδηγίας αυτής και εκεί αναφέρει διάφορα ζητήματα. Πάντως, η άλλη πτυχή, ο άλλος βραχίωνας της ομάδας εμπειρογνωμόνων, αναφέρθηκα σε αυτό στην αρχή, επικεντρώθηκε κυρίως στο εξή θέμα, κατά πόσο η οδηγία αυτή προσαρμόζεται ως έχει τώρα στις ε, challenges, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την αγγλική λέξη, στις δυσκολίες, στις προκλήσεις ε, που έχουμε από την τεχνητή νοημοσύνη και κατά πόσο πρέπει να υποβληθούν κάποιες ε, προτάσεις για αλλαγές. Δεν υπάρχει τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το παρόν, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Επιτροπής. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω από αυτού. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Γκονζάλης όχι. Α, α δεν θέλετε το λόγο. Καλώ. Ωραία, τότε νομίζω τελειώσαμε αυτό το θέμα. Mm. Α, ε, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο κύριο Σενμάιερ, μας έδωσε πάρα πολλές λεπτομέρειες και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα συνεχιστεί αυτή η ανταλλαγή απόψε. Θα σας προσκαλέσουμε και πάλι μέσα στους επόμενους μήνες για να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας. Είναι, θα είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συνάντηση. Ωραία. Καλώς. Οπότε τελειώσαμε με αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι ψηφοφορίες. Πρώτη ψηφοφορία. Νομική βάση, άρθρο 40. Πρόκειται πληροφορίες ε, ηλεκτρονικές για τις μεταφορές, εμπορικές μεταφορές. Μας έχουν ζητηθεί τρεις ε, γνωμοδοτήσεις βάσει του άρθρου 42, σύμφωνα με τον κανονισμό. Ε, ναι, παρακαλώ, όσοι αποχωρείτε από την αίθουσα, παρακαλώ ησύχως. Γιατί αυτοί που ψηφίζουν πρέπει να καταλάβουν τι ψηφίζουν. Συμφωνεί. Λοιπόν, η Λίμπε και η Τρανς έχουν ζητήσει. Η κυρία Ρομπέρτη θέλει να ζητήσει το λόγο πριν προχωρήσουμε. Παρακαλώ. Α, όχι κύριε Ρομπέρτη. Όχι. Ωραία, η πρώτη γνωμοδότηση έχει να κάνει με την νομική βάση όσον αφορά την ακτοφυλακή και τα σύνορα. Τι δεν λειτουργεί. εξετάζει θέμα αυθεντικότητας εγγράφων που προσφέρονται ηλεκτρονικά. Θα ψηφίσουμε λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Παρακαλώ ησυχία για να μπορούμε να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Είπα, η πρώτη ψηφοφορία έχει να κάνει με την γνωμοδότηση επί της νομικής βάσης όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Εκτοφυλακή για ε, παραπημένα ευθυντικά έγγραφα online, FADO, το σύστημα αυτό. Πρόκειται για την ε, κοινή δράση του Συμβουλίου 98700JHA και είναι κάτι που ζητήθηκε από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ψηφίζουμε λοιπόν. Μπορείτε να ψηφίσετε. Shall we take this vote by... Πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. I apologize, the system is not working. Δεν λειτουργεί το σύστημα από ό,τι φαίνεται. Sorry, it was working just now. Yes, yes. Okay. <laughs> So we now hope that we can open the vote. Ωραία, τώρα μάλλον μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Εντάξει, λειτουργεί. Καλώς. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Δεύτερη γνωμοδότηση. Γνωμοδότηση επί της νομικής βάσεως για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πληροφορίες εμπορικών μεταφορών. Πρόκειται για το 2018 κάθετος 0140. Μπορείτε να ψηφίσετε. Άλλος ένας. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Και το επόμενο πρόκειται για την γνωμοδότηση νομική βάση αποφάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά τη Γερμανία και την Ιταλία να μπορούν να τροποποιήσουν κάποιες διμερείς συμφωνίες ε, που έχουν για τις οδικές μεταφορές με την Ελβετία 2019-01-07 και 2019-01-08. Ψηφίζουμε. Πέρα στις φοφορίες. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Σημείο 8. Προσαρμογή κάποιων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης για τη χρήση κανονιστικών διαδικασιών με έλεγχο βάσει του άρθρου 290. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά με πλειοψηφία των μελών μας. Χρειαζόμαστε δηλαδή 13 ψήφους υπέρ για να περάσει. Ψηφίζουμε λοιπόν. Τέλος. Σημείο Νομική πράξη για κανονιστικές διαδικασίες, ε, πάλι από το άρθρο 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάλι ψηφίζουμε για να ξεκινήσουμε διοργανικό διάλογο. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σημείο 10 δράσεις για την προστασία των ε, συλλογικών αποζημιώσεων καταναλωτών. Πάλι για να μπούμε σε διοργανικό διάλογο. Ε, ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της προφορίας. Εγκρίθηκε. Σημείο 11. Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη-μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικέ και εμπορικέ υποθέσεις. Και πάλι μπαίνουμε σε διαπραγματεύσεις διοργανικές. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σημείο 12. Συνεργασία μεταξύ των δικαστήριων των κρατών μελών κατά την διεξαγωγή αποδείξεων κτλ. Πάλι μπαίνουμε σε διαπραγματεύσεις. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Σημείο 13. Αναφορά σχετικά με τις συμβατικές ρήτρες που χρησιμοποιούν μη εμπορικές οντότητες συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων δημιουργού. Πρόκειται για μία επιστολή Θέλει κανείς να πάρει το λόγο πριν ψηφίσουμε. Όχι. Α, ο κύριος Μπρέια, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την πρόταση αυτή απάντηση, γιατί δεν αντιμετωπίζει τις ελλείψεις, τις σοβαρές αδυναμίες των καθεστώτων, στα οποία αναφέρεται ο αναφέρον και γι' αυτό εμείς θα καταψηφίσουμε. Ευχαριστούμε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω απλώ να πάρω το λόγο για να συγχαρώ την Προεδρία για την απάντηση που πιστεύω ότι είναι πολύ ε, συνολική, που δεν επιδέχεται καμία ερμηνεία ε, στραβή όσον αφορά την πραγματικότητα. Γιατί μπορεί κανείς να έχει ό,τι δεν θέλει και να χειρίζει τα θέματα με σλόγγαν και ιδεολογία, αλλά νομικά τα πράγματα είναι έτσι όπως ακριβώς πολύ απτά τα αναφέρει η απάντηση. Οπότε συγχαρητήρια για αυτή τη συνθετική ικανότητα. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ κύριε Πρέη. Επιτρέψτε μου να απαντήσω σε αυτό. Φυσικά. Σωστά είπατε ότι πρόκειται για το νομικό καθεστώ, αλλά ακριβώ αυτό το νομικό καθεστώ θέλει να τροποποιήσει ο αναφέρον. Και η επιστολή λέει τι υπάρχει και λέει ότι δεν πρέπει να αλλάξει. Νομίζω ότι εντάξει είχαμε αρκετά ανταλλαγή απόψεων, αν δεν θέλει κανένας άλλος να πει κάτι διαφορετικό. Ωραία, ψηφίζουμε, παρακαλώ, ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Σημείο 14. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία. Αναδιατύπωση. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της προφορίας. Ευχαριστώ. Και τέλος σημείο 15. Πρόκειται για την απαλλαγή 2018. Ο κύριος Λεμπρετό είναι εισηγητής. Θέλει μήπως να πει κάτι ο κύριος Λεμπρετό. Παρακαλώ. Όχι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα έχουμε πει για το θέμα αυτό. Είναι περιττό. Ναι, ψηφίσαμε επί μακρό για τις τροπολογίες, πράγματι. Ένα παραγράφος 2α. Ψηφίζουμε. Πέρασε τις φοφορίες. Πέρασε η τροπολογία. Επόμενη τροπολογία, τροπολογία 2. Μπορείτε να ψηφίσετε παρακαλώ, η τροπολογία 2. μπορειτε να ψηφισετε παρακαλω τροπολογια 2 περασε εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 4. 5 ψηφίσατε πέρας 6 Πέρας. Εγκρίνεται. 7. αυτό τίποτα. Τέλος. Εγκρίνεται 8. Τέλος προφορίας. Απορρίπτεται 9. Τέλος. Εγκρίνεται. 10. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 11. Α, όχι, πάμε στη 12. 12. 13 και 14 μαζί. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Δε... Τροπολογία. Α, η 15 καταπίπτει. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος, της πρότασης. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ. Τώρα, περνάμε και κλεισμένο το θυρών για να κάνουμε την τελευταία ψηφοφορία. Λίγα λεπτά θα κρατήσει. Δύο λεπτά. Απλώς θα βγαίνουμε από το web streaming κλείνει το web streaming, η αναμετάδοση στο διαδίκτυο δηλαδή, για να ψηφίσουμε και κλεισμένο το αθυρόν. Ναι,